Meine Damen und Καλωσορίζω κυρίες και κύριοι στην σημερινή μας πρωινή συνεδρίαση. Εχθές δυστυχώς δεν ήμουν σε θέση να προσέλθω στη συνεδρίασή μας διότι μέσω της Κυριακής ε, το, το βράδυ είχα αποκλίνει λίγο λόγω των εκλογών. Περνάμε στο σημείο 8 της ημερησίας διάταξης. Ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Στοκχόλμης. Η συγητής είναι ο συνάδελφός μας κύριος Μπισέπ. Κύριε συγητά, έχετε κάποιες παρατηρήσεις να κάνετε. Τι λέτε. Δεν έχετε κάποιες παρατηρήσεις. Περνάμε λοιπόν τώρα στην ψήφιση. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 1, παρακαλώ. Κατά θα ελέγξουμε λοιπόν. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Υποθέτω ότι εγκρίθηκε. Πέρα Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Απορρίφθηκε όμως παρόλα αυτά. Συμβιβασμός 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε στην τροπολογία 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε 7 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε 8 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Ίδιες πλειοψηφίες πάντα. Και περνάμε τώρα στην τροπολογία 11 υπέρ απορρίφθηκε η 8, η 9 υπέρ, 9 κατά αποχές εγκρίθηκε. Να ελέγξουμε όμως, ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, σαφές το αποτέλεσμα. 9 λοιπόν. 9. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 9. Πέρας ψηφοφορίας με 22 υπέρ 42 εναντίον απορρίφθηκε. Ποιος είναι υπέρ της 10 κατά άποχες απορρίφθηκε. 11 υπέρ κατά εσ. Θα ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 11. Ή 11 είναι που ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε 36 ψήφοι υπέρ, 28 εναντίον, 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 13 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίθηκε. Υποθέτω. Να ελέγξουμε ή συμφωνείτε ότι εγκρίθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν. Ήταν ασαφές το αποτέλεσμα. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε και περνάμε τώρα στον συμβιβασμό 2 υπέρ κατά αποχές. Ο συμβιβασμός απορρίφθηκε νομίζω. Θα ελέγξουμε όμως. Ψηφίζουμε τον συμβιβασμό ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την τροπολογία 17. Πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε με 28 υπέρ 35 εναντίον. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 22 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 27 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 28 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε. Υποθέτω απορρίφθηκε, αλλά θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. 45 υπέρ 18 εναντίον. Εγκρίθηκε. 29 με προφορική τροποποίηση υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 35 σε τμήματα. Το πρώτο τμήμα, όσοι είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Θα ελέγξουμε για το πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε το σύνολο του κειμένου. Τέλος ψηφοφορίας. Με 54 ψήφους υπέρ 11 εναντίον εγκρίθηκε. Θερμά συγχαρητήρια. Και περνάμε τώρα στην έκθεση για τη βιομηχανική πολιτική, για το διάστημα, τον χώρο του διαστήματος. Ποιο θα ήταν καλύτερα ενδεδειγμένο και κατάλληλο για αυτό το θέμα από την κυρία Κρόνμπεκ. Έχετε κυρία Κρόνμπεκ κάποιες παρατηρήσεις να κάνετε. Όχι, δεν είσαστε. Α, στην τροχιά στο διάστημα. Εντάξει, ωραία. Περνάμε τώρα και ψηφίζουμε το κείμενο. Συμβιβασμός 1, υπέρ εγκρίνεται. Συμβιβασμό 2 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχέ εγκρίθηκε. 9 υπέρ κατά αποχέ εγκρίθηκε. 10 υπέρ κα, κατά απόχέ εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε στον συμβιβασμό 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε το κείμενο, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας με 52 υπέρ 6 κατά 5 αποχές εγκρίθηκε θα αποστείλουμε ένα μήνυμα με τον ασύρματο στην κυρία εισηγήτρια. Και περνάμε τώρα στην κατάσταση στην περιοχή του Σαχέρ την κατάσταση για τα δικαιώματα του ανθρώπου εκεί. Η είναι ο κύριος Τάνοκ. Έχετε κάτι να μας πείτε εισαγωγικά κύριε Τάνοκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για το μήκος και την περιπλοκότητα του κατάλογου ψηφοφορία. Ήταν πολύ πολλωμένη συζήτηση που μας διέρεσε. Πολλά από τα προβλήματα που αφορούν τα, τα θέματα της Δυτικής ε, Σαχάρας, του Σαχέλ, είναι πολύ προβληματικά. Ζητώ την υπομονή σας και την ανοχή σας. Ελπίζω ότι αυτό που θα προκύψει θα είναι μια ισορροπημένη έκθεση. Ξέρετε ότι λόγω της περιπλοκότητας κάθε λέξη μετράει. Είναι περίπλοκη συζήτηση, περίπλοκο το κείμενο, υπάρχουν πολλές τροπολογίες, πολλές συμβιβαστικές τροπολογίες, αλλά ελπίζω το αποτέλεσμα να είναι αρκετά ικανοποιητικό από όλε τι πλευρέ για να περάσει το κείμενο στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου για περαιτέρω αλλαγές είμαι σίγουρος. I think here it's a record record. 36 compromises. Έχουμε 36 συμβαστικές τροπολογίες. Είναι ρεκόρ αυτό. Πάντα έχουμε μπροστά μας νέες προκλήσεις. Kompromiss 1 dafür. Συμβιβασμός 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 90 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 95 υπέρ. Κατά. Και πάλι. 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 101 με ναι. το κείμενο όπως αναφέρεται συμπληρωματικά υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Τώρα περνάμε στο συμβιβασμό 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 104 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 108 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 109 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Εκα... Αυτή ήταν η 109, συμβιβασμός 6 τώρα. Α, η 110 πιο πάνω, ναι, 110 τώρα, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 6, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 116, υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 117. Να ελέγξουμε, να ελέγξουμε την 116. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Abstimmung ist ψηφοφορίας λειτουργήσε η τάση της ε, ανωτικής αριστεράς και του ΕΛΚ, εγκρίθηκε αυτή. 117 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 118 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 119 υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκε. 120 υπέρ, κατά αποχές. Ασαφές το αποτέλεσμα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Νομίζω απορρίφθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. Με 41 ψήφους υπέρ, εναντί 24 εναντίον εγκρίθηκε. 121 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 122 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. Συμβασμός 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 127 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 130 σε τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ μέχρι εκεί που λέει ο given policy μιας δεδομένης πολιτικής υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Για το δεύτερο τμήμα τώρα υπέρ κατά εγκρίθηκε. 132 τροπολογία υπέρ κατά θα ελέγξουμε ψηφίζουμε την 132 ηλεκτρονικά άρχεται τέλος ψηφοφορίας αποτέλεσμα 34 υπέρ 32 εναντίον εγκρίθηκε συμβασμός 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβασμός 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 139 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 140 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε μετά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 Εγκρίθηκε η 159 λέει ο πρόεδρο. Πέρα ψηφοφορία εν πάση περιπτώσει. 35 υπέρ 30 εναντίον εγκρίθηκε. 160 υπέρ κατά αποχέ εγκρίθηκε. 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 163 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβασμός 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 166 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 167 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Εντάξει. 167 λοιπόν. Άρχι, πέρας ψηφοφορίας. 26 υπέρ 38 εναντίον. Απορρίφθηκε. 168 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 168 ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. με 28 υπέρ 37 εναντίον απορρίφθηκε. 169 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 175 υπέρ. Κατά ελέγχουμε ηλεκτρονικά. 175. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα. 29 υπέρ 37 εναντίον απορρίφθηκε. 176 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 100... καταπίπτει άλλη. 178 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 181 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 182 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε αυτό ισχύει όσον αφορά τον τύπο και όσον αναφέρεται την επισήμανση το 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 184 υπέρ κατά αποχές Απορρίφθηκε. Αλλά θα ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 184. Τέλος ψηφοφορίας. Με 37 υπέρ 28 εναντίον εγκρίθηκε. 188 τροπολογία υπέρ. Κατά. Επειδή συμμετείχα εγώ δηλαδή υπερψηφίστηκε, εγκρίθηκε. 189 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 190 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 191 υπέρ. Κατά αποχές. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 191 ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα. 36 υπέρ, 29 εναντίον εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 18. Α, η 192 πρώτα, υπέρ. 192 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 196 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. 197 υπέρ κατά εγκρίθηκε να ελέγξουμε διαμαρτύρονται εντάξει τέλος ψηφοφορίας 35 υπέρ 30 εναντίον εγκρίθηκε η τροπολογία λυπάμαι Η 197 ήταν αυτή, έτσι. Τώρα πάμε στην 198. Ηλεκτρονικά. Αν εγκριθεί, να ενταχθεί χωρίς να υπάρχουν επικαλύψεις. Ποιοι είναι υπέρ της 198 λοιπόν. Κατά. Απόχες εγκρίθηκε. 199 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 200 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 201 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 204 υπέρ κατά 204 και πάλι ποιοι είναι υπέρ Κατά. Εγκρίθηκε. 205 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 205 ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. 29 υπέρ 30 εναντίον απορρίφθηκε. Συμβιβασμός 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 209 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 210-211 για το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Για ποια χώρα πρόκειται εκεί, τι είναι, για τις παράλληλες αυτές τροπολογίες που έχουμε. Ποια πρεσβεία θα μπορούσε να στείλει θετικές ειδήσει. 213 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 212 όχι 214 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 215 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 216 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 217 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 218 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 219 υπέρ κατά θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 219 ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. 39 υπέρ 26 εναντίον εγκρίθηκε. 220 υπέρ. Κατά. Α, εγκρίθηκε. 221 υπέρ. Όχι. 221 η 219 απορρίφθηκε λέει ο πρόεδρος. Εγκρίθηκε. Α, αφού εγκρίθηκε η 219, 223 τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 224 υπέρ. ελέγξουμε την 223 ηλεκτρονικά. Τροπολογία 223 λοιπόν. Τέλος ψηφοφορίας. Με 26 ψήφους υπέρ 38 εναντίον απορρίφθηκε η τροπολογία αυτή. Τροπολογία 224 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 225 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 21 υπέρ. Κατά εγκρίθηκε. 229 υπέρ κατά απορρίφθηκε. 230 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 231 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 232 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 233 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 236 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 237 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Σύμβασμος 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 200, 240 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβασμός 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 243 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβασμός 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 248 υπέρ 248 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. 249 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 252 υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ της 252 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. Πάμε τώρα στην τροπολογία 253 υπέρ. 253 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. 40 υπέρ, 23 εναντίον. Εγκρίθηκε. Αλλά δεν με πιστεύει κανείς όταν το λέω. 254 τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 258 υπέρ. Κατά αποχές. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. 38-26 εγκρίθηκε. 261 υπέρ. ...261 υπέρ... ...κατά... ...αποχές... ...θα ελέγξουμε λοιπόν ηλεκτρονικά... τελος πληροφορια ψηφοφορίας. 36-29 εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα, ποια ήταν αυτή, η 259 τώρα, έτσι. Ωραία, ποιοι είναι υπέρ 259. Κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 260 υπέρ. Κατά, αποχές απορρίφθηκε. Συμβασμός 27 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Συντροπολογία 266 υπέρ. Κατά. 266 εντάξει υπέρ. Και πάλι 266 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 266. Πιστεύω όμως ότι απορρίφθηκε. Τέλος ψηφοφόρειας. 29 υπέρ 36 εναντίον. Απορρίφθηκε. 263 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 200... απορρίφθηκε αυτή η 271 και περνάμε τώρα στην 267 267 υπέρ κατά Αποχέσα. απορρίφθηκε 268 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 272 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Οι σοσιαλιστές υπερψηφίζουν, οι άλλοι καταψηφίζουν. Στην τροπολογία αντρικένε δηλαδή, έτσι. Τέλος ψηφοφορίας. 36 υπέρ 23 εναντίον. Εγκρίθηκε. Είχα πει ότι είχε εγκριθεί. 273, όχι, καταπίπτει. 274 υπέρ. 273. 273 τώρα. Υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 273. Τέλος ψηφοφορίας. Κρίμα που δεν είναι η Βερονίκη εδώ. Θα λέγει ότι δεν είχε λειτουργήσει η συσκευή της. Λοιπόν. 274 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε με την προφορική τροποποίηση. Πάντα όπως έχει επισημανθεί στο κείμενο, όπως αναφέρεται στο κείμενο. Η τροπολογία συμβαστική 28. Συμβαστική 28 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 278 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. 282 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε τροπολογίες 283, 84, 85 Ταυτόσημες υπέρ αυτών κατά αποχές. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε αυτές τις τροπολογίες ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα Πέρας ψηφοφορίας είπα. 34 υπέρ, 30 εναντίον εγκρίθηκαν οι τροπολογίες αυτές. ...294 υπέρ... ...κατά... ...αποχές απορρίφθηκε... ...295 υπέρ... ...κατά... ...αποχές απορρίφθηκε... ...296 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 297 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 298 σε δύο τμήματα και με μια προφορική τροποποίηση κιόλας ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τρίτο τμήμα. Έχουμε και ένα τρίτο τμήμα, μάλιστα. Remaining munitions, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 299 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 300 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 301 υπέρ. Κατά, αποχές απορρίφθηκε. Συμβιβασμός 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε στην τροπολογία 303 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Περνάμε στην τροπολογία 309 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 310 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 311 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Θα ελέγξουμε λοιπόν, μάλιστα. Τέλος ψηφοφορίας. 45 υπέρ, 16 εναντίον. Εγκρίθηκε. Οι λομπίστες ε, με το μήνυμα το οποίο αποστέλλεται ήταν ιδιαίτερα επιτυχής. 314 τώρα. υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 315 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 316 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 318 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 317 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 320 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 319 σε δύο τμήματα. Ποιοι είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία Μάιερ, υπέρ, κατά, αποχές. Η 321 είναι, έτσι, όχι η Μάιερ, η 321, συγγνώμη, μάλιστα. 321 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 322 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Να ελέγξουμε, ελέγχουμε λοιπόν, 322, μα είχε Παρακαλώ, εν πάση περιπτώσει, τους συναδέρφους να σηκώνουν ξεκάθαρα τα χέρια τους και να συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Είναι πολύ μικρή η διαφορά πολλές φορές και αν κάποιοι δεν ε, ψηφίζουν τότε δεν μπορούμε να δούμε ποιο είναι πραγματικά το αποτέλεσμα. Εγκρίθηκε λοιπόν, μάλιστα, εγκρίθηκε αυτή. Συμβιβασμός 30, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Περνάμε στην 327 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 327 ηλεκτρονικά. <coughs> Πέρας ψηφοφορίας. 31 υπέρ, 30 εναντίον εγκρίθηκε. 328 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Αλλά θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 300. Ή συμφωνείτε ότι απορρίφθηκε. Έστω ελέγχουμε. «23 υπέρ 40 εναντίον απορρίφθηκε, 329 υπέρ, 329 υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκε, 330 υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκε. 332 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 333 υπέρ. 332 λέτε αυτήν. Ωραία. Πέρας ψηφοφορία στην 332. 25 υπέρ 38 εναντίον. Απορρίφθηκε. 333 τώρα. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 334 υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε τη 334 ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. 30 υπέρ, 31 εναντίον. Απορρίφθηκε. 335 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 336 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβιβασμός 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 331. Μόνο το πρώτο τμήμα όμως εδώ. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 337 υπέρ κατά αποχές Ένα τρίτο των μελών μόνο συμμετείχαν στην ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ της 337 παρακαλώ. Κατά άποχες εγκρίθηκε. Τι είπατε. Ήταν σαφές το αποτέλεσμα όμως. Πέρας ψηφοφορία σε πάση περιπτώσει. 38 υπέρ 24 εναντίον. Εγκρίθηκε λοιπόν. Μάλιστα. 341 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Περνάμε τώρα στις αιτιολογικές σκέψεις. έχουμε μεγάλο τμήμα λυρικών παρατηρήσεων, οπότε μπορεί να είναι και κάποια οδύε. Τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 26 υπέρ με ένα μπάρο δύο τριγώνια 25-26 από κοινού πέρας ψηφοφορίας. 23 υπέρ, 36 εναντίον απορρίφθηκαν. 27 υπέρ, κατά, αποχές. Δεν πρόσεχα, δεν είδα το αποτέλεσμα. 27 υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε, ψηφίζουμε την 27.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 28 υπέρ 33 εναντίον. Απορρίφθηκε. Η 33 είπαμε είναι γλωσσική μορφή Η 34 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. «35 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε». Συμβιβασμός 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τοπολογία 40 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 41, 42 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 43 υπέρ κατά εγκρίθηκε. 44 υπέρ Η 43 ήταν η προηγούμενη, έτσι. ψηφοφορίας. 31 υπέρ 28 εναντίον εγκρίθηκε. 44 υπέρ κατά αποχές. Φαίνεται ότι απορρίφθηκε, αλλά εντάξει, πάμε στις 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 34 είπε 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 54 υπέρ 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός 36 για την 59. Πέρας ψηφοφορίας για την 59. Θα ελέγξουμε λοιπόν δύο φορές, με διπλό έλεγχο έστω. Συμβιβασμός 36 τώρα, υπέρ. 36 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε τώρα στην τροπολογία 63. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 64 υπέρ. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. 67-68 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκαν. 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 70 σε δύο τμήματα απορρίφθηκε είπα εγκρίθηκε ενώ απορρίφθηκε απορρίφθηκε λοιπόν η 69 70 υπέρ Έχουμε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά. Θα ελέγξουμε λοιπόν το δεύτερο τμήμα. Δεύτερο τμήμα της 70. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Εγώ πιστεύω ότι είχε εγκριθεί. Τέλος ψηφοφορίας. 34 υπέρ 25 κατά εγκρίθηκε. Τρίτο τμήμα τώρα υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 73 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Πού είναι οι υπόλοιποι της ομάδας. 20 δεν έχουν ψηφίσει ακόμα. Τι γίνεται. 73. 73. Πέρας ψηφοφορίας επί της 73. 32 υπέρ 30 εναντίον. Εγκρίθηκε. Σωστό. 74 τώρα υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Εν πάση περιπτώσει ελέγχουμε και πάλι. Η 74 δεν είναι που ελέγχουμε. Ωραία. Απορρίφθηκε. Σωστό. Λοιπόν, παρακαλώ τώρα σε αυτόν τον τελευταίο γύρο να σηκώνετε τα χέρια και να ψηφίζετε ή να συμμετέχετε στην ψηφοφορία. Εν μέρει οι φιλελεύθεροι δεν συμμετέχουν καν. Παρότι ήταν δική τους κιόλας η τροπολογία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. 75. Α, ποιοι είναι υπέρ της 75. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 76 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε θα λέγα. Η 75 απορρίφθηκε, απορρίφθηκε και η 76. 77 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 78 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 79 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβασμός 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε τώρα στην τροπολογία 84 σε τρία τμήματα. Ποιοι είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Για το δεύτερο τμήμα τώρα, υπέρ, εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα, ψηφίσαμε πριν το πρώτο τμήμα. Τώρα ψηφίζουμε το δεύτερο, έτσι. Ποιοι είναι υπέρ του δεύτερου τμήματος. Κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά, αποχές απορρίφθηκε. Ποιος είναι αυτός που ζητά διαρκώς έλεγχο και έλεγχο, τσεκ. Τέλος ψηφοφορίας. Όχι, όχι ακόμα, δεν έχουμε τελειώσει με την ψηφοφορία. Τώρα, πέρας ψηφοφορίας. 26 υπέρ εναντίον. Απορρίφθηκε. Η 85 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Πάμε τώρα στην τροπολογία. 2, 2 σωστό. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Μπορούμε να τις πάρουμε μέχρι την 11 όλες μαζί. από 6 έως 11 από κοινού. Ομού. Μέχρι τη 10. Εντάξει. Από την 6 έως την 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκαν. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 13. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 14 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 16 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε τώρα στις τροπολογίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Αν ψηφίσουμε τις ΔΕΒΕ της Επιτροπής Ανάπτυξης τις 10 για την 10. Ποιοι είναι υπέρ λοιπόν την 10. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Για τις υπόλοιπες τοπολογίες της ΔΕΒΕ. Όλες τις υπόλοιπες υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκαν. Πάμε στην Επιτροπή Γυναικών τώρα. Τοπολογίες Επιτροπής Γυναικών. συμφωνήσαμε Έχω διαφορετικό κατάλογο. Έχω Ψηφίσαμε ξεχωριστά την ΤΕΒΕ 10. Για την 6, 7, 8 έχω διαφορετικά πρόσημα. Πήγαμε τώρα πιο γρήγορα. Εμείς ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Ρώτησα τι θα επιθυμούσατε. Τώρα περνάμε στην Επιτροπή Γυναικών. Ένα. Τροπολογία 1. Τροπολογία Επιτροπής Γυναικών 1. Έχουμε διαφορετικές τροπολογίες μπορούμε να πάρουμε την, από την 1 έως, τις, έως ε, την 9 από κοινού. Όχι, δεν συμφωνείτε, δεν είναι δυνατόν. Θα τις πάρουμε επιμέρους τις τροπολογίες εξειδικευμένα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι εδώ πρόεδρος, εντάξει και δεν κάνουν άλλοι παρατηρήσεις. Εντάξει, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, γίνονται εδώ διάφορες παρατηρήσεις, οδηγούν στο χάος. Τροπολογία γυναικών 1, φαμ 1, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. ΦΑΜ 2 έως ΦΑΜ 9. Ούτε και αυτό το δέχεστε. Λοιπόν, κάθε μία ξεχωριστά. Τροπολογία ΦΑΜ 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 4 υπέρ. Κα... Κατά αποχές εγκρίθηκε. 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 10 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 11 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε εντάξει φαμ 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 13 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 14 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 15 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ψηφίζουμε τη 15 ηλεκτρονικά πέρας ψηφοφορίας 35 υπέρ, 27 εναντίον, εγκρίθηκε. Τροπολογία 16 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 18 υπέρ, κατά Με μερική συμμετοχή του ΕΡΚ εγκρίθηκε η 18, εν πάση περιπτώσει, 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 26 υπέρ κατά λέει ο πρόεδρος υπέρ και πάλι επαναλαμβάνουμε 26 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε 27 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε 29 υπέρ. Κατά αποχές. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 29 ηλεκτρονικά. Εγκρίθηκε λοιπόν. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 36 υπέρ. Πώς είπατε εσείς.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 αποχές εγκρίθηκε 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε πάμε τώρα στην ηλεκτρονική τελική ψηφοφορία στο σύνολο του κειμένου άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά τέλος ψηφοφορίας Με 46 ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον, 13 αποχές εγκρίθηκε. Θερμά συγχαρητήρια. Επιτρέψτε μου τώρα δύο παρατηρήσεις για αυτό. Παρακαλώ και πάλι να ξαναδούμε με αυτές τις ταυτόσιμες ε, τροπολογίες που όλο και περισσότερο κατατίθενται τέτοιες παράλληλες ταυτόσιμες ε, τροπολογίες. Όταν έχουμε τέτοιες ταυτόσιμες που δεν έχουν συζητηθεί και αναλυθεί, τότε μπορεί να υποθέτει κανείς ότι ε, έχουμε ταυτόσιμη, ας το πω έτσι, πηγή προέλευσης ε, για το 1 τρίτο αυτόν. Στο διευρυμένο Προεδρείο πρέπει να το δούμε. Ένας τρίτος φαίνεται, ένας τρίτος με συγχωρείτε συντάσσει αυτές τις τροπολογίες και δεν ανταποκρίνεται στην αξιοπρέπεια και κύρος του Ευρωκοινοβουλίου να έχουμε τέτοιου είδους προσέγγιση, τέτοιου είδους διαδικασία από τρίτους να συντάσσονται. Επιπλέον πρέπει μια συναρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή να υποβάλει 41 τροπολογίες. Είναι υπερβολικά πολλές, είναι δυσανάλογο αυτό. Out of proportion, υπερβολικά δυσανάλογο. Και στο μέλλον θα πρέπει μια τέτοια κατάσταση να την εξετάσουμε εκ του σύνεγγυς, να δούμε τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Και περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη που είναι και κλεισμένων των θυρών όμως, πράγματι και κλεισμένων των θυρών